Okay, colleagues, if Συνάδελφοι, έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Έχουμε την Επίτροπο, έχουμε πολλά. Θα ήθελα να σας αναφέρω τι, καν, τι είπαν οι συντονιστές αποφάσισαν δύο εκθέσεις να γίνουν. Μία από το ΕΛΚ και μία από τους σοσιαλιστάς. Η λεγόμενη Connecting Europe Facility πρέπει να τύχει της άδεια για να γραφτεί έκθεση από τους προέδρους, από τη διάσκεψη των προέδρων. Θα σας αναφέρω νεότερα λοιπόν. Έχουμε την ημερήσια διάταξη, Διδέχεστε. Τότε περνάμε στο 3, ανταλλαγή απόψεων με τον Μακλέιν, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Θα μιλήσει για 10-15 λεπτά, μετά θα γίνει πρώτος γύρος σε ρωτήσεων από συντονιστέ και συντονίστριες και μετά δεύτερος γύρος για όλους και όλες. Και μετά Επίτροπος Χέντγκαρντ. Λοιπόν, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ή, ή η διευθύντρια, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, έχετε μπροστά σας την έκθεση για τις πρασινότερες μεταφορές. και για τον ενδεικτικό μηχανισμό πληροφόρησης για τις μεταφορές και το περιβάλλον. Για δεύτερη φορά ερχοπανίζομαι ενώπιόν σας, γιατί το πρόγραμμα αυτό συζητιέται σε πολλές φάσεις. Κατά κάποιον τρόπο είναι καλά τα νέα, δηλαδή η τελευταία έκθεση λέει ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα περιβαλλοντικός Μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών καταρτήσαμε τον λεγόμενο οδικό χάρτη των μεταφορών που είναι νομίζω για σας κάτι το πολύ χρήσιμο για να ενημερωθείτε. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία του 9 κυρίως. Η παρουσίασή μου λοιπόν θα αναφέρει πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να πάμε και με τι ταχύτητα. Γενικά σημειώνουμε, παρατηρούμε πρόοδο και βελτιώσεις. Θα μιλήσω λοιπόν για τις εκπομπές, την ενέργεια, το θόρυβο και την βιοπικιλότητα γιατί αυτά τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι εχθές άρχισε να συγγράφεται και η έκθεση για την ποιότητα του αέρος. Πάντως οι εκπομπές για όλους τους ρήπους έπεσαν το 9. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην ύφεση. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δυστυχώς βλέπουμε όμως ότι η ποιότητα του αέρος έχει χειροτερέψει το διοξίδιο του αζότου ιδιαίτερα. διότι μπορεί να δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα και οι οριακές τιμές έχουν ξεπεραστεί σε 41% των σταθμών μέτρησης. Η κατανάλωση ενεργείας για τις μεταφορές συνεχώς αυξανόταν τα τελευταία χρόνια, αλλά μεταξύ 8 και 9 η γενική η ζήτηση ενεργείας έπεσε κατά 4%. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει γιατί άμα λήξει η ύφεση θα αυξηθεί η κατανάλωση ενεργείας. Η χορύπανση σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι ακόμη εκτίθενται σε ηχορύπανση από αυτοκίνητα και φορτηγά. Για πολλούς λόγους συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό γιατί υπάρχουν αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανης που δεν αφορούν μόνο το θόρυβο, προβλήματα ύπνου κλπ. Επίσης οι, επιστημονικοί, οι επιστήμονες δείχνουν ότι μπορεί η χορύπανση μέσω του διαταραγμένου ύπνου να διαταράξει και την ανάπτυξη των παιδών. Ο θόρυβος λοιπόν και η χορύπανση είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Όπως ξέρουμε οι μεταφορές πάντοτε είχαν επιπτώσεις και στη βιοπικιλότητα οι αυτοκινητόδρομοι και τα λοιπά. Και βλέπουμε μάλιστα ότι ακόμα και μόνο στο Βέλγιο πολύ μεγάλο ποσοστό του εδάφους καλύπτεται από τσιμέντο. Το 30% βέβαια μόνο του ευρωπαϊκού εδάφους καλύπτεται από δρόμους, αλλά και αυτό πολύ είναι. Γιατί χάνεται βιοπικιλότητα και μέχρι το 20 πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα, πού θέλουμε να πάμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές βελτιώσεις, μερικές οφείλονται στην ύφεση, αλλά υπάρχουν και θετικά στοιχεία και πρέπει να δούμε με τι κίνητρα, τι κίνητρα πρέπει να εφαρμόσουμε. Οι τιμές των καυσίμων έχουν πολύ ψηλές τιμές, αλλά μόνο 15% υψηλότερες ήταν το 9 σε σύγκριση με το 80. Δεν είναι λοιπόν η τιμή των καυσίμων το κυριότερο κριτήριο για τις επιλογές που πρέπει να κάνουμε για τις μεταφορές. Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να δούμε ότι έχουν επιτέλους καθοριστεί καθολική σφαιρικοί στόχοι για τις μεταφορές που δίνουν μία ένδειξη στους πολιτικούς και σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για τις επιλογές που πρέπει να κάνουν. Γενικά δεν, το θέμα δεν είναι μόνο η στόχη, είναι και η αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών. Σας μίλησα για τους ρήπους του αέρος. Η δομοθεσία για τις εκπομπές δεν διορθώνει πάντοτε τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη διαφορά μεταξύ των στόχων που θέτουμε εμείς στην ομοθεσία και των αποτελεσμάτων στην ποιότητα του αέρα. Δεν έχουμε καταλήξει σε καθαρισμό του αέρος λοιπόν. Υπάρχουν ακόμη πολλά, πολλοί ρήποι που δεν τους έχουμε λάβει υπόψη. Τώρα, μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Η Κομισιόν προτείνει να μειωθεί η εκπομπή των εκπομπών θερμοκηπίου, όπως ξέρετε, 60%, κατά 60% μέχρι το 50% και το 90%. Το 2009 οι μεταφορές και οι θαλάσσιες και οι χερσές ε, ε, δημιούργησαν σχεδόν το 25% των εκπομπών. Επομένως, δυστυχώς, κυρίως οι οδικές μεταφορές, χερσαίες μεταφορές, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για τις εκπομπές αυτές. Θα χρειαστούν λοιπόν τεράστιες περικοπές. Δεύτερος στόχος για τις μεταφορές επιβατών, για τις συγκοινωνίες. Έχουν και εδώ σημαντικέ αυξήσεις σημειωθεί, ιδίως στις αεροπορικές μεταφορές αλλά και στις οδικές. Φυσικά με την ύφεση βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή πτώση αλλά σχεδόν ασήμαντη. Οι περισσότερες μεταφορές γίνονται οδικός με αυτοκίνητα ιδιωτικά και με με λεωφορεία αλλά κυρίως με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Τι προτείνει λοιπόν η Κομισιόν να κινηθούμε προς ένα αποτελεσματικότερο σύστημα μεταφορών. Το 30% των οδικών μεταφορών μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους τρόπους όπως σιδηροδρομικές. Και τι λέμε άρα, ότι οι μεταφορές εμπορευμάτων έχουν πέσει σε μεγάλο βαθμό για αποστάσεις μικρότερες των 300 χιλιόμετρων, αλλά και αυτό οφείλεται στην ύφεση. Οι οδικές μεταφορές δυστυχώς κυριάρχησαν έναντι των σιδηροδρομικών και άλλων. Κυρίως λοιπόν οδικά γίνονται ακόμη οι μεταφορές τα καύσιμα με λιγότερη εκπομπή διοξιδίου είναι ένα ακόμη μία λύση που συζητάμε και μέχρι το 50 πρέπει κατά 40% να μειωθούν οι εκπομπές από καύσιμα κατά 40% ή και 50%. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας That we continue to work on. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Τέλος, η πρότασή μας να μειωθούν οι μεταφορές με τα συμβατικά αυτοκίνητα ή με τα αυτοκίνητα που συμβατικά καύσιμα είναι επίσης μια πρόταση που ζητάμε τα εναλλακτικά καύσιμα υπάρχουν ήδη και αρχίζουν να χρησιμοποιούνται. Τα περισσότερα τέτοια αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα LPG, λίγα είναι μόνο τα ηλεκτρικά. Η κυκλοφορία λεωφορείων με αέριο έχει αυξηθεί και αυτή και το ποσοστό και άλλων λεωφορείων με αναλλακτικά καύσιμα υπάρχει αλλά δεν είναι πολύ ψηλό. Εμείς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε για τα αιτήματά σας για τη χρησιμοποίηση περισσότερων αυτοκινήτων με λιγότερες εκπομπές. Τα νέα αυτά αυτοκίνητα το 10 ήταν κατά ένα πέμπτο αποτελεσματικότερα από ό,τι την περασμένη δεκαετία. Τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε μια τελική ενημέρωση για τα καινούργια αυτά αυτοκίνητα αλλά δεν θα δούμε εκεί ποιο είναι ο μέσος όρος εκπομπής διοξιδίου του άνθρακο από αυτοκίνητα. Γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ των δοκιμών των πειραματικών αυτοκινήτων και της πραγματικής τους χρήσης. Στην έκθεση βλέπετε, θα δείτε ότι υπάρχουν γραφικές παραστάσεις που δείχνουμε το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να το πετύχουμε. Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτά. Ελπίζουμε λοιπόν να συνεχίσει να σημειώνεται πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς και ότι θα καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα πιο συγκεκριμένο όπου θα μπορούμε να σας πούμε τι συμβαίνει γενικότερα όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών αλλά και γύρω από αυτόν. Όλες οι παράμετροι που αφορούν την αύξηση εκπομπών γιατί βλέπουμε ότι είναι πολλοί οι στόχοι και το θέμα είναι μπορούμε να τους πετύχουμε όλους ή πρέπει να διαλέξουμε πρώτα και να προτιμήσουμε ορισμένους. Αυτά. Σας κατευχαριστούμε. Κύριε Μακλέιντ. Τώρα ο κύριος Γκρός από το ΕΛΚ. ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ο θέλω στην Ιταλία. Έχουμε... Είχαμε ελάχιστο χρόνο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε την έκθεση. Η πρώτη ερώτηση αφορά στα 300 χιλιόμετρα για τα οποία μιλάει η Κομισιόν. Έχετε στοιχεία κατά τα οποία μπορείτε να μας μιλήσετε για τις μεμονωμένες χώρες και κατά δεύτερον, η ενεργειακή κατανάλωση, την οποία υπολογίζεται και περιγράφεται ανά είδος μεταφοράς, είναι η κατανάλωση ενέργειας μόνο για τη χρήση και την ε, κίνηση του ε, οχήματος ή και για την παραγωγή του. Και τρίτη ερώτηση σε ό,τι αφορά ε, την αυτιλιακή πολιτική, η διαφορά μεταξύ ε, βορρά κοινό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και κάποιο καιρό κάποιοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα ότι φυσικά το θείο στα λιμάνια είναι πολύ επικίνδυνο για την ε, ανθρώπινη υγεία και στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά θα μπορούσε να είχε θετική επίδραση στο κλίμα. Θα μπορούσατε να τοποθετηθείτε. Αυτή ήταν η τρίτη ερώτηση και τώρα η τέταρτη ερώτηση το e-mobility τις επόμενες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά πολλά από την ηλεκτρονική αυτή κινητικότητα. Ε, από πού θα προέλθει όμως αυτή η ενέργεια, αυτό το ρεύμα, μήπως αυτή η ηλεκτρονική κινητικότητα θα είναι πιο επιβλαβής από ότι η παραδοσιακή ε, παραγωγή ενέργειας. Και τελευταία ερώτηση, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ αμα, οχήματος και χρήστη, επιβάτη, να πούμε ε, ότι το εξής, μιλάτε για ε, λεωφορεία, για παράδειγμα, τα οποία είναι απόλυτα γεμισμένα. Αυτές ήταν οι πέντε ερωτήσεις που είχα να κάνω. Thank Σας ευχαριστώ για το S&D, για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Αλκαντράουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίασή σας, κυρία Μαγκλέιτ. Μιλήσατε για την Λευκή Βίβλο, μεταξύ άλλων, όπου αναφέρεται ότι στην πολιτική μας ε, η πολιτική μεταφορών ε, θα έχει αυξηθεί κατά 80% μέχρι το 2050. Άρα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Συμφωνώ μιλήσατε για κάποιες ε, στοχοθεσίες. Αλλά αναρωτιέμαι το εξή, σε ό,τι αφορά το μείγμα των μέτρων που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο, για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πώς αξιολογείτε τις προτάσεις εκείνες, ποιες θεωρείτε ότι είναι ουσιώδεις, σημαντικές, ποιες θα έπρεπε να θέσουμε ως προτεραιότητες για να αλλάξουμε πραγματικά κάτι σε ό,τι αφορά το τοπίο των μεταφορών. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ξέρετε ότι πολλές από τις προτάσεις αυτές θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, η συζήτηση για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Μεταφορών στο Κοινοβούλιο και στην Οδηγία για την Ραβινιέτα και για τον ε, τομέα των οδικών μεταφορών. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να θέσω ως ερώτηση. Δεύτερη ερώταση που συνδέεται και με την ερώτηση του κ. Γκρόση για τα 300 χιλιόμετρα. Φυσικά αυτό έχει να κάνει με ε, μεταφορές ε, μεγάλης απόστασης, αλλά ξέρουμε ότι οι μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα, η μεγαλύτερη ε, επιβάρυνση είτε από η χορύπανση ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει στις μικρές αποστάσεις και εκεί μπορεί να είναι μεγάλο το όφελος όταν ρυθμίσουμε τα πράγματα καλύτερα. Και εδώ λοιπόν η ίδια ερώτηση. Βράχει στι σχετικά. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να ειναι μεγαλο το όφελο οταν ρυθμισουμε τα πραγματα καλυτερα και εδω λοιπον η ιδια ερωτηση βραχει προθεσμα σχετικα τι πιστευετε οτι θα πρεπει να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ωραίο είναι να θέτουμε στόχους για το 2050. Απέχει πολύ ακόμα, αλλά θα πρέπει και βράχει πρόθεσμα να ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Ποια είναι τα, οι, οι γρήγορες αυτές οι λύσεις που θα προτιμήσετε για να πετύχετε. Αυτά. Thank you, Mrs. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μακλέιτ για την παρουσίασή της. Και εγώ έχω παρατηρήσεις και ερωτήσεις να κάνω. Καταρχάς, μία ερώτηση γιατί θα πρέπει ασφαλώς πρώτα να ε, μελετήσουμε την παρουσίαση αυτή. Τα ευφυή e συστήματα μεταφορών ε, θα ελεγχθούν ως προς την αποτετικότητά τη, γιατί ιδιαίτερα στις αστικές μεταφορές, όσο πιο καλή είναι η μεταφορά στον αυτοκινητόδρομο, τόσο πιο λίγα είναι τα ατυχήματα και τόσο πιο αποτελεσματικές είναι οι μεταφορές, τόσο πιο χαμηλές είναι και οι εκπομπές που εκλείονται. Έχουν γίνει σχετικές μελέτες, έχετε αριθμητικά στοιχεία να μας παρουσιάσετε. Κατά δεύτερον, να συμφωνήσω και εγώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκρός σε ό,τι αφορά τις εκπομπές θείου στα πλοία. Αυτό μας απασχολεί, όχι μόνο επειδή θέλουμε να τις μειώσουμε, αλλά εγώ που είμαι από την Βόρεια Γερμανία, οι επιτρεπόμενες εκπομπές είναι 0,1%. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει μετακύληση στον αστικό τομέα. Τι μπορείτε να μας πείτε όμως για το θέμα αυτό. Μήπως υπάρχει τεχνολογία σκράμπε που θα μπορούσε να ε, ε, εφαρμοστεί το LNG από ένα θέμα, το ευρωποιημένο αέριο, το οποίο θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις ε, στον τομέα των μεταφορών μέσω θαλάσσης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά το όριο των 300 χιλιόμετρων που προτάθηκε, ασχοληθήκαμε πριν από λίγο με τη Λευκή Βίβλο και θα συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Γκρό. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι τοπικέ ιδιαιτερότητε. Φυσικά μπορούμε να πούμε 300 χιλιόμετρα είναι το όριο και να θέσουμε και ένα σχετικό ποσοστό για την ε, μεταφορά μέσω οδών, μέσω σιδηροδρομικών ε, ε, οδών, αλλά φυσικά άμα δεν υπάρχει θάλασσα, τι νόημα έχει να θέσουμε αυτή την προϋπόθεση. Άρα θα πρέπει να θέσουμε αυτό το τοπικό χαρακτήρα. Ένα τελευταίο θέμα, το οποίο δεν έχει αναφερθεί ακόμα, για την αστική μεταφορά. Πολλά μπορούν να επιτευχθούν, γιατί όντω νομίζω ότι πάνω από 50% των ε, ιδιωτικών οχημάτων εμ, ε, κάνουν αποστάσεις μικρής εμβέλειας στον αστικό τομέα. Πολλά μπορούν να βελτιωθούν λοιπόν. Να προταθεί, για παράδειγμα, ηλεκτρονικά ποδήλατα ε, με μέτρα δημοσίων μεταφορών. Μπορεί να μην είναι πανάκια αυτά τα ηλεκτρονικά ποδήλατα, αλλά μπορεί να σημειώσουν μία πρόοδο. Και να τονίσουν, αν θέλετε, και τον αθλητικό χαρακτήρα ανθρώπων που κατά τα άλλα δεν έχουν ευκαιρία να κουνηθούν ιδιαίτερα, να ασκηθούν ιδιαίτερα στη δουλειά τους, στην καθημερινή του ζωή. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Σκράμερ για τους πράσινους. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, Διευθύντρια για την έκθεση. Και όλα αυτά αποτελούν επιπρόσθετες αξίες, επιπρόσθετες τιμές. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε δύο λόγια για το χρηματικό σκέλος. Ε, είναι περίεργης ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει φόρος κυροζήνης ε, και άλλοι ε, ευνοούνται ενώ άλλοι δεν ευνοούνται. 60% των ε, κονδυλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνε στο δρόμο και 20% μόνο στους σιδηροδρόμους. Και επίση χρηματοδοτούνται λάθο προγράμματα. Υπάρχει συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, για μια νέα σύνθεση συνδρομική μεταξύ Στουτγκάρντε και Ούλμη και χρειάζεται νέα λοιπόν ε, ε, τέτοια ε, γραμμή ενώ υπάρχει η παλιά γραμμή η οποία δεν ενδείκνεται όμω για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Και η καινούργια όμω γραμμή δεν μπορεί να εξυπηρετεί εμπορεύματα. Άρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Και αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αποδεχόμαστε πλέον. Δεν κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την χορύπανση παρόμοια είναι τα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να μειωθεί η χορύπανση. Αλλά με αντίστοιχο πρόγραμμα 4,5 δισεκατομμυρίων για τα εμπορεύματα θα μπορούσαμε να πετύχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Άρα δεν χρησιμοποιούν το σωστό τρόπο τα χρήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη χρηματική διάσταση, να πούμε ότι και τα μεγάλα προγράμματα ευνοούνται. Τα μεγάλα προγράμματα όμως ε, πότε θα πραγματοποιηθούν δεν μας ενδιαφέρει σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Φυσικά θα πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το ρεύμα, αλλά καθοριστικό είναι και η όλη ε, αλυσίδα της παραγωγής, της χρήσης και της ανακύκλωσης. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα είναι καλύτερα από τα παραδοσιακά, αλλά το Γερμανικό Υπουργείο είπε ότι θα, μειώσουμε κατά 25% τις εκπομπές αερίων αν ε, τα εφαρμόσουμε και μιλήσατε και για την κατανάλωση αναέκταση. Να σας πω ότι η γερμανική κυβέρνηση θέλει μέχρι το 2020 να μειώσει, θέλει να μειώσει την ε, θέλει το Γερμανικό Υπουργείο να μειώσει κατά 30 εκτάρια μέχρι το 2020 την ε, κατανάλωση αυτή ανά επιφάνεια. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Και να σας πω ότι κάθε αυτοκίνητο ακόμη στη Γερμανία ε, επιδοτείται ακόμα με 500 ευρώ. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην έχω αυτοκίνητο, αλλά πληρώνω για το αυτοκίνητο του γείτονά μου. Μπορείτε να μας πείτε αν ισχύει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τελευταίο σημείο, μιλήσατε με τη διαφορά, για τη διαφορά μεταξύ της ε, χρήσης και της ε, παραγωγής και της κατανάλωσης. Μας είπατε ότι πολλές φορές γίνονται διάφορα κόλπα. Αλλά τι χρησιμοποιείτε εσείς για να κάνετε, να καταπολεμήσετε αυτές τις διαφορές. Μάλιστα, αν θα θέλετε να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, κύριε Μακλέιτ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λεγοντα το εξή. Απαντώντας συνδυαστικά για τα 300 χιλιόμετρα, νομίζω ότι ειλικρινά ως είδος φιλοδοξίας είναι κάτι το απόλυτα εύλογο, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά θίξατε ότι υπάρχουν περιφερειακές διαφορές και αυτές θα μπορούσαν να καταστήσουν την εφαρμογή α... αδύνατη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν την χωρική διάσταση και σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα, γιατί σαφώς υπάρχουν θέματα βιοπικιλότητας για το πώς θα επιλύσουμε τα διάφορα είδη μεταφορών και ίσως να μην υπάρχει μία λύση για όλους. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μία καλή εξέταση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή χρήση. Έχουμε πληροφορίες ανά χώρα και ανά τομέα μεταφορών. Υπάρχει και ένα πίνακας πίσω, στο πίσω μέρο τη έκθεση. αλλά αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι οικοδομέ ε, ο κατασκευαστικό κλάδο. Στην παρούσα φάση δεν συμπεριλαμβάνεται όλος ο κύκλος ζωής ε, των οχημάτων. Άρα πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εξετάσουμε ποια είναι τα υλικά. Και σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, και σε ό,τι αφορά άλλους τομείς της κατασκευής ενός οχήματος. Αλλά σαφώς, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά θέματα που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Άρα, δεν είναι απλή, απλώς ο υπολογισμός για την ενεργειακή κατανάλωση. Αλλά γίνεται σχετικό έργο στην παρούσα φάση και νομίζω ότι θα μας ενδιέφερε να επανέλθουμε στο σημείο αυτό στο μέλλον. Τώρα, για το θείο. Φυσικά υπάρχουν ε, ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ βορρά και νότου, αλλά θα πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό από περιβαλλοντικής άποψης ε, και να πούμε το εξή, ότι υπάρχει πιστοποίηση για τις εκπομπές, αλλά το θείο εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά μας και επηρεάζει διάφορα οικοσυστήματα. Βλέπουμε ότι επηρεάζει και τα ύδατα, αλλά βλέπουμε ότι το διοξίδιο του θείου και η έκθεση στο θείο στις αστικές περιοχές είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε συνδυασμό με το όζον, ε, σχηματίζει ένα ανθραντιφόρο μείγμα και ανακύπτει θέμα ανθρώπινης υγείας σε ό,τι αφορά το διοξίδιο του θείου. Άρα δεν πρόκειται για κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι «Α, το αντιμετωπίσαμε, πάει τελείωση». Υπάρχει λοιπόν πολύ, υπάρχουν πολλοί λόγοι υπολογίζοντας και το κόστος των ζημιών που έχει υπολογίσει η υπηρεσία μας και όλα αυτά καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το θείο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και στις αστικές ε, περιοχές, γιατί πραγματικά είναι σχετικά τα επίπεδα, αλλά και πάλι το θέμα αυτό άπτεται και της ε, έκθεσης ε, για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Από πού προέρχεται το ηλεκτρικό για την ηλεκτρονική κινητικότητα. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ διαφορετική ικανότητα εξέταση σήμερα της πρόσβασης των χωρών στην, στην ε, ανανεούμενη ενέργεια. Οι χώρες θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για, την, ε, για τις ανακτικές πηγές ενέργειας. Και νομίζω ότι αυτό θα καλύψει και τις ανάγκες της ηλεκτρονικής κινητικότητας μέσα στο αστικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι γίνεται φυσικά και για τις μεγάλες αποστάσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά μέσα στις πόλεις νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε και θα μπορέσουμε να καλύψουμε στο μέλλον τις ανάγκες αυτές. Ίσως δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε οι ικανότητες αυτές, αλλά πρόκειται να γίνει αυτό στο μέλλον. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με τις επιδοτήσεις, αλλά από πλευρά ενέργειας πιο πολύ. Και έχουμε υποδείξει ότι είναι σημαντικό το θέμα των επιδοτήσεων στον τομέα μεταφορών. Θα ξαναξεκινήσουμε μια σχετική μελέτη, τις οποίες ονομάζουμε μελέτη για τις ε, επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, αλλά τις αναφέρουμε απλά ως επιδοτήσεις. Αναμφίβολα αυτό το θέμα παραμένει στο τραπέζι και το κατά πόσον ε, συγκαταλέγεται στον οδικό χάρτη αποδοτικότητα πόρων ή όχι, σίγουρα θα πρέπει να συζητηθεί και σίγουρα θα πρέπει να συζητηθεί για να είναι αποτελεσματική η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίσιμο αυτό για μας. Κατά πόσον αυτό θα οδηγήσει σε δημοσιονομική και φορολογική μεταρρύθμιση, αυτό εξαρτάται από τις πρωτεύουσε. Αλλά για να σας δώσω κάποια στοιχεία. Στην παρούσα φάση συζητάμε με διάφορα κράτη-μέλη, τα οποία σοβαρά εξετάζουν ενδεχόμενη φορολογική μεταρρύθμιση για να μετατοπιστεί το βάρος της φορολόγησης ε, προς τους πόρους. Είναι πάρα πολύ έντονη η δυναμική και στις συζητήσεις μας και στην διαδικασία και είμαι βέβαιη ότι θα ξέρετε από τις χώρες σας να θα ξέρετε από τις χώρες ότι θα υπάρξει ανάγκη να εξεταστεί η φορολογική βάση, καθότι αλλάζει και η σύνθεση του πληθυσμού και άρα το θέμα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους υπουργούς οικονομίας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο οι μεταφορές, αλλά και η συλλογή εσόδων σε εθνικό επίπεδο. Για την ε, διάκριση των μεταφορών ανατομέα. Ναι, περιλαμβάνονται αυτά στην έκθεση και υπάρχει ανάλυση κατά χώρα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια χώρα στην οποία ο κόσμος να ταξιδεύει πιο πολύ με λεωφορεία ιδιαίτερα ή με άλλους τρόπους. Τώρα, ε, με ρωτήσατε κατά πόσον βασιζόμαστε ε, και κάνουμε υπολογισμούς βάσει λεωφορείων ή οχημάτων που είναι απόλυτα γεμισμένα. Όχι. Υπάρχει ένα ποσοστό για το μείγμα τώρα των μέτρων και πρακτικέ προτάσει. Νομίζω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι συνεκτική είναι ενδεκτική για αυτά που κάναμε στο πακέτο για την ενέργεια, που υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Προτείνουμε μεταξύ άλλων να δούμε πόσο ρεαλιστικά είναι όλα τα μέτρα και κατά πόσο σε τελική ανάλυση μας παρέχουν κίνητρα επενδύσεων σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα, το 2012 σκοπεύουμε να εξετάσουμε τη δέσμη όλων των στόχων που έχουν τεθεί, είτε από τον τομέα του περιβάλλοντας, της ενέργειας των μεταφορών και από τους δικούς μας τομείς, περιλαμβάνεται και η γεωργία, για να δούμε πώς συνδυάζονται και κατά πόσον υπάρχουν ε, τομείς πραγματικά που το ένα μέτρο αντιβαίνει στο άλλο. Δεν έχω μία απάντηση να σας δώσω, αλλά κατά το επόμενο έτος θα έχουμε μία πολύ καλύτερη ιδέα για το πώς συνδυάζονται τα μέτρα αυτά. Για την ηχορύπανση, έχετε δίκιο. Υπάρχουν κάποια βραχυπρόθεσμα ωφέλη. Αν με ρωτούσατε σήμερα, επί τι θα πρέπει να θέσουμε ως στόχο, νομίζω ότι η ηχορύπανση αποτελεί ασφαλώς ένα ενδυμικό πρόβλημα, το οποίο πλήττει τους πάντες. Εκατοντάδες εκατομμύρια πλήττονται από επίπεδα ηχορύπανσης που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται. Και αυτή η ηχορύπανση η χαμηλής, ε, χαμηλού επίπεδου. Τώρα, κατά πόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα, αυτό, το θέμα αυτό μέσω σχεδιασμού, μέσω σχηματισμού ζωνών, ε, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και φυσικά θα πρέπει να επανέλθω στο κατά πόσο έχουμε λάβει υπόψη ε, ευφύης ιδέες για τον σχεδιασμό. Ναι, αλλά ένα βασικό θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε και να προσαρμόσουμε ήδη οι υφιστάμενες δομές στον αστικό τομέα. Υπάρχουν πόλεις όπως η Βαρκελόνη για παράδειγμα όπου εξετάζεται τέτοιο ενδεχόμενο μέσω ηλεκτρονικών ποντήλατων για παράδειγμα και άλλων συστημάτων για τον κύκλο ελέγχου. Στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης υπάρχει ένας πίνακας ε, συνοπτικός, ο οποίος και πάλι εξετάζει μεταξύ, της διαφορές μεταξύ των εκπομπών και του κύκλου ελέγχου. Γιατί άμα αναφέρεται γιατί ασφαλώς και υπάρχουν διαφορές. Στο μείγμα αυτών μέτρων θα πρέπει να κοιτάξουμε τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού αποτελέσματος και του θεωρητικού αποτελέσματος, το οποίο μπορεί θεωρητικά να θέτει ένα πολύ καλό παράδειγμα, αλλά στην πραγματικότητα να μην μας βοηθάει ιδιαίτερα για τη χρήση τώρα των γεών. Τη χρήση του εδάφους βλέπουμε ότι η φυστάμενη δομή μεταφορών επηρεάζει ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό περιβάλλον για την ε, απορρόφηση μολυντών μέσω της γεωργίας, μέσω του εδάφους κτλ. Και άρα το πλαφόν που έχουμε, το, τα επίπεδα που παρατηρούνται σήμερα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και αυτό προκύπτει και από την ανάλυση hot που καταδεικνύει ότι υπάρχουν μέρη στην Ευρώπη που δεν θα έπρεπε να οικοδομούνται άλλα κτίρια, για παράδειγμα, ή άλλοι δρόμοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ανώτατα όρια, τα οποία καθιστούν α, κάποιες περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες και που απειλούν και τον ίδιο τον πληθυσμό τελικά. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Σκούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Μακλέιτ για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Στην ατζέντα του 2020 και στη Λευκή Βίβλο για την ε, κινητικότητα του μέλλοντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά την προσαρμογή της χρήσης ενέργειας και το όριο των 300 χιλιόμετρων παίζει ένα ρόλο. Τώρα κατά πόσον αυτά είναι εφαρμόσιμα ή κατά πόσον θα αντιδράσει διαφορετικά η οικονομία δεν μπορούμε να το προβλέψουμε από τώρα, θεωρώ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξή. Όλες οι δραστηριότητε οι οποίες γίνονται σήμερα σε ό,τι αφορά την μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα στον τομέα της, του, των μεταφορών, θα πρέπει να συντονιστούν όλες αυτές οι ενέργειες. Η εκπομπή, για παράδειγμα, αντεξοδίου του άνθρακα για μικρά οχήματα έχει ρυθμιστεί. Συζητάμε τεχνική ανανέωση και νέες μηχανές καύσης. Πολλά μέτρα συζητάμε, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούν. Το καθοριστικό είναι ότι χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σαφή για τους μεμονωμένους ε, κλάδους ε, μεταφοράς. Πόση ενέργεια καταναλώνεται ανά τόνο, ανά χιλιόμετρο, ανά ναυτικό μίλι. Υπήρξε θετική εξέλιξη με τα μέτρα μας τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τον καταναλωτή, για να έχουμε μία βάση επί της οποίας μπορούμε να συνεχίσουμε την κατάρτιση της στρατηγικής μας. Να πούμε ότι για παράδειγμα στην ε, μεταφορά μέσω θάλασσας ε, υπήρξε αύξηση της ε, κατανάλωσης ενέργειας κατά 27% για παράδειγμα. Και να ξέρουμε πού κινούμαστε. Θα πρέπει να υπάρχει όμως μια ακριβής ανάλυση. Και επίσης, το είπε και ο κύριος Γκρός, πόσο μπορούμε να πετύχουμε μείωση του θείου χωρίς να, υπάρχουμε, να υπάρχει μεταφορά σε άλλο είδος μεταφορών. Θα πρέπει να κρατήσουμε τις τιμές αυτές του 0,1 ή μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον δεν είναι ρεαλιστικές αυτές οι τιμές. Και αυτό που είναι πολύ βασικό, επειδή οι πόροι και τα ρηκτά καύσιμα μειώνονται, θα πρέπει να έχουμε τεχνικές καινοτομίες, θα πρέπει να τις ε, ενισχύσουμε και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί κοινό καθήκον και της ε, οικονομίας αλλά και της ε, Ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία μου για όλα αυτά τα στοιχεία και τους αριθμούς. Αλλά διαπιστώνω με όλες τις συζητήσεις ε, που έχουμε κάνει εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο, ακούγοντας εσάς δηλαδή και τους άλλους, διαπιστώνω ότι είμαστε όλοι εδώ στο κοινοβούλιο σχιζοφρενείς. Δηλαδή έχουμε τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να ε, αξιοποιήσουμε την ε, ζήτηση, αλλά μετά μιλάμε και για την προσφορά και στην περίπτωση των και το, το θέμα δηλαδή ε, της ε, βελτίωσης ε, της προσφοράς με, αυτές τις, με αυτή τη ζήτηση για για δρόμους αναπνοής, άρα ενισχύουμε τις μεταφορές, δηλαδή έχουμε low cost για τις αεροπορικές εταιρείες, μειώνουμε ε, τους αεροπορικούς ναύλους και εγώ ήμουν υπουργό μεταφορών. Σίγουρα καταλήγουμε σε ορισμένους συμβιβασμούς. Αλλά πρέπει εδώ να το παραδεχτούμε ότι όλοι είμαστε σχιζοφρενείς, λέμε ένα πράγμα και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Θα πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο σε θέμα για θέματα χωροταξίες, για την κατάργηση του αυτοκινήτου και το ποδήλατο στην πόλη, εγώ σίγουρα δεν είμαι κατά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. αυτό είναι, αυτά είναι τα κατεπήγοντα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά το μοντέλο ολόκληρο της παραγωγής, της κατανάλωσης, ε, να μπορέσουμε να εργαστούμε και στην ζήτηση των μεταφορών, όχι μόνο στην ε, προσφορά και στη διαχείριση των τιμών. Αυτό είναι το βασικό θέμα, δηλαδή αυτό που θέλουν να καταστήσουν ε, τη μεταφορά πολιτικό ζήτημα και όχι μόνο οικονομικό ε, και σίγουρα οι μεταφορές έχουν και αυτή την πτυχή, αλλά κύριε μου, για το θέμα της ε, ζήτησης. Θα υποβάλλετε προτάσεις πέρα δηλαδή και από τα δικά σας ε, παιδί αρμοδιοτήτων, δηλαδή πέρα από το περιβάλλον υπάρχει το θέμα της χωροταξίας, υπάρχει το θέμα της οικονομίας. Δηλαδή βγαίνουμε ευθύ αμέσω ε, από το περιβαλλοντικό μοντέλο, φτάνουμε στο γενικότερο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δημιουργεί περισσό, ανάγκη για περισσότερες μεταφορές, για περισσότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος κλπ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να πω και εγώ μια δυο λόγια. Πρώτον, νομίζω ότι οι χρήστες και οι επιχειρήσεις των μεταφορών καλώς ή κακώς θεωρούν ότι οι μεταφορείς και οι μεταφερόμενοι θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι για την καταστροφή του περιβάλλοντος και αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό. Στη σελίδα 43 της έκθεσής σας μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς συναδέλφους το γεγονός ότι στην τρίτη παράγραφο εκεί λέτε ότι την περασμένη δεκαετία αυξήθηκε η ζήτηση σιδηροδρομικών μεταφορών ενώ η ανταγωνιστικότητα τους υποβοηθήθηκε από το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρόμων. Μήπως εδώ κάτι δεν καταλάβαμε, διότι <clears throat> εμείς δεν πιστεύουμε ότι έχει ανοίξει η αγορά των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Ίσα ίσα συζητήσαμε πάρα πολλές ώρες ζητώντας από την Κομισιόν να κάνει περισσότερα για να ανοίξει την αγορά των σιδηροδρόμων, των σιδηροδρομικών μεταφορών δηλαδή. Άρα εδώ διαφωνώ. Και πιο κάτω λέτε ότι 25% των συνδρομικών μεταφορών υψηλή ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 25% μόνο, αλλά το υπόλοιπο 75% των συμβατικών μεταφορών τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι καν ηλεκτρικό σε αυτές οι συνδρομικές μεταφορές είναι με ντίζελ. Και γι' αυτό σας ρωτάω, όταν γράφετε τέτοιες εκθέσεις ελέγχετε καθόλου αν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Και από εδώ τίθεται προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Θα μπορούσε κανείς να γράψει ολόκληρο ντοκτορά. Μπορεί κανείς να σχεδιάσει την αύξηση αυτών μεταφορών χωρίς να μειώσει την κινητικότητα. Γιατί έτσι είπατε. Και εδώ το ερώτημα για τους χρήστες ιδίως και τους οδηγούς που πηγαίνουν με το αυτοκίνητο 100 μέτρα για να, βάλουν τα παιδιά στο, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο γιατί φοβούνται τους κακοποιούς. Τι θα σημαίνει για αυτούς η μείωση της κινητικότητας, μία μείωση της κινητικότητας. Όσο για τις αεροπορικές μεταφορές και την φορολόγηση των καυσίμων της, Δεν είμαι βέβαιος ότι εσείς υποστηρίζετε ή όχι αυτή τη φορολόγηση, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι φρονείτε. Γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι δεν μπορεί μόνο η Ευρώπη να κάνει τέτοια φορολόγηση, να αυξήσει το κόστος, δηλαδή μόνο εκείνοι και οι άλλοι να εφελούνται. Το ίδιο ισχύει και για τη βενζίνη των αυτοκινήτων. Πιστεύετε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση σημαίνει ότι πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω να φορολογηθούν παραπάνω τα ορυκτά καύσιμα Πιστεύετε επίσης ότι υπάρχει θέμα να πείσουμε τον κόσμο ότι ότι πρέπει η φορολόγηση των καυσίμων να εφαρμοστεί για να υπάρξει βιώσιμη για να υπάρξουν βιώσιμες μεταφορές. Πολλοί υπουργοί έχω ακούσει να το υποστηρίζουν αυτό, αλλά ως υπουργοί μεταφορών αλλά όταν γίνονται υπουργοί οικονομικών το απορρίπτουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε αν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι για να υπάρξουν βιώσιμες μεταφορές χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όχι να πούμε, όχι δεν έχετε το δικαίωμα να πάρετε το αυτοκίνητό σας για διακοπές ή να το αεροπλάνο. Ορίστε κύριε Μαγκλέιντ. Ας αρχίσω με τη χιζοφρένεια. Αυτό που βλέπουμε όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά σε όλους τους πόρους, είναι αυτό το πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης που πρέπει να εξισορροπηθεί με κάποιο λογικότερο τρόπο. Θα έλεγα ότι η διαχείριση μέσω της αγοράς όταν δεν αναγνωρίζετε ότι υπάρχει σπάνις των πόρων είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει σπάνις που είναι κάτι που χειρίζεται καλύτερα από όλα η αγορά. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα μέτρα που προτείνονται μερικές φορές φαίνονται ως τιμωρία για τους χρήστες και εδώ μπορεί να παίξει ρόλο η φορολογική μεταρρύθμιση. Πρέπει να δοθεί και κάποια επιβράβευση, κάποιο κίνητρο δηλαδή, στους μηχανισμούς που προωθούν τη βιώσιμη μεταφορά. Τώρα το κατά πόσον το σωστό που θα επιβραβεύεται γίνεται και με φορολογία είναι ένα ερώτημα που τίθεται στο παρελθόν Ήδη οι χρήστες υπέστησαν την ύφεση και η δυνατότητα να πηγαίνουν διακοπές σε μακρινούς τόπους είναι κάτι που περιορίστηκε. Αλλά τι εννοούμε εμείς κινητικότητα του 21ου αιώνα. Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο λεπτομεριακά. Παρά το γεγονός ότι η ύφεση φέρνει τα πράγματα κυρίως στα δημοσιονομικά. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο είναι η ασφάλεια και η υγεία. Άρα μπορούμε να πούμε με ισχυρά επιχειρήματα ότι η επένδυση σε καθαρές μεταφορές, εναλλακτικές μεταφορές είναι κάτι που θα ωφελήσει τους τομείς αυτούς, την υγεία και την ασφάλεια. Αλλά αυτά βέβαια πρέπει να προκύψουν από ένα κοινωνικό αίτημα, να εξηγηθούν οι επιπτώσεις που θα είχε η συνέχιση της τωρινής κατάστασης. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης της ενέργειας. Αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το κύριο είναι να ξέρει ο κόσμος αν βοηθιέται έτσι στην καθημερινή του ζωή και αν μπορεί να το πληρώσει το βιώσιμο τρόπο. Αυτό ισχύει και για τον τομέα των υδάτων. Δεν θεωρείται μεν βασικό δικαίωμα, αλλά σχεδόν η κινητικότητα. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί κανείς να πληρώσει το κόστος της και τις επιπτώσεις της. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για κινητικότητα και πώς θα μπορούσε αυτή να εφαρμοστεί καλύτερα σε αστικό περιβάλλον, στις πόλεις δηλαδή. Το θέμα δεν είναι απλώς η περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά ο διάλογος με τους κατοίκους των πόλεων. αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα στατιστικά στοιχεία και κριτήρια για τις πόλεις, δηλαδή τα μέρη όπου ζει το 70-75% του πληθυσμού, θα μπορούσαμε να έχουμε σοβαρά επιχειρήματα για την ηχορύπανση, την ποιότητα του αέρα κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για μία σαφή αλλαγή της επιχειρηματολογίας, να τονίσουμε περισσότερο πού μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αυτό πιο αποτελεσματικοί στις πόλεις μπορούμε να είμαστε. Όσο για τις μακρών αποστάσεων μεταφορές, εκεί πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα και κατά πόσον θα μιλήσουμε για το σιδηρόδρομο, τις μεταφορές εμπορευμάτων ή τις ποτάμιες μεταφορές. Βλέπουμε όμως τις συζητήσεις των φορολογικών μεταρρυθμίσεων ότι αν ο κόσμος δει ότι πληρώνει περισσότερα για κάτι όμως που του αποφέρει κάτι στην υγεία και την ασφάλεια, θα το καταλάβει. Αλλά πρέπει και για την ενέργεια και για το νερό όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα απαρχαιωμένων υποδομών και χρειάζονται νέες επενδύσεις, να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους επιχειρήματα με προτεραιότητες, να δούμε δηλαδή ποιες υποδομές πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα γιατί θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί πρέπει το πρόβλημα να το λύσουμε επιγόντως. Το 2020 είναι μόνο 9 χρόνια μετά. Δεν αρκεί ο χρόνος αυτός για να αλλάξει το τύπος αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιούμε μέχρι τότε. Πρέπει να δούμε πώς συνδυάζονται όλοι μαζί οι στόχοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πιο πιστικό και για τους πολίτες. Να μπορούσαμε να τους πούμε, ορίστε, τα σοβαρά επιχειρήματα τα θετικά που θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση, αν και μπορεί να σημαίνει υψηλότερο κόστος. Δεν αρκεί να πει κανεί όχι είναι ακριβά αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακλέιτ, και για την παρουσίαση της έκθεσης και για την απάντηση στα σχόλια και στις ερωτήσεις των βουλευτών. Να ρωτήσω λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής ε, να σας ζητήσω να εκφράσουμε την ε, εκτίμησή μας με τον συνήθι τρόπο. Είχα ε, σαφείς οδηγίες να αφήσω την κυρία Μαγκλέιτ να φύγει γιατί έχει και ένα τρένο να προλάβει στις 10.30. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Okay. Thank you. Okay, colleagues, we Μάλιστα, συνάδελφοι, και έχουμε την Επίτροπο μαζί μας ήδη. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, πέντε λεπτών, μην απομακρυνθείτε και όταν έρθει η Επίτροπος Χέντικαρτ θα ξεκινήσουμε πάρα αυτά. Okay, colleagues, can I reconvene the meeting and, and welcome Commissioner Connie Hedegaard. Χαιρετίζω την Επίτροπο Κόνι Χέντεγκαρντ για την δράση για το περιβάλλον, για το κλίμα. Έχουμε καμιά ώρα. Θα σας δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο για την παρουσίασή σας περίπου δεκάλεπτη και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν ενδιαφέροντα σχόλια οι συνάδελφοι. Ορίστε κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν τέτοιο διάλογο. Έχω συναντήσει μερικά από τα ε, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής σας, αλλά όχι με το σύνολό της. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό για μένα αυτό που συζητάτε και για τις μεταφορές που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος και ευθύνεται για ένα τέταρτο όλων των εκπομπών. Οι οδικές μεταφορές είναι η κύρια πηγή, 70% των εκπομπών από μεταφορές. Όπως μάλλον ξέρετε, ο δικός μας χάρτης για μία ανταγωνιστική χαμηλών εκπομπών οικονομία μέχρι το 50 δείχνει ότι οι άλλων ειδών μεταφορές μειώνονται από το 90 και μετά στους υπόλοιπους τομείς εκτός από τις μεταφορές όπου όλα αυξάνονται. Άρα στον τομέα αυτό είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα πράγματα όσα έχουν θα χρειαστούν μειώσεις από όλους τους παράγοντες του τομέα αν θέλουμε ως Ένωση να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομπών. Η μείωσή τους είναι λοιπόν ουσιαστικό μέρος της κλιματολογικής μας στρατηγικής. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Επιτροπή Μεταφορών θέλει να μειωθούν οι εκπομπές με τόσο φιλόδοξο τρόπο όπως το εξέφρασε στην Λευκή Βίβλο. Στη δική μας Λευκή Βίβλο είχαμε θέσει ορισμένους ενδεικτικούς στόχους και ενδιάμεσους το 2020, 30, 40 Ιδίω η μείωση των εκπομπών διοξιδίου κατά 20% μέχρι το 30. Αυτό είναι χαμηλότερο από τους στόχους για άλλους τομείς, ότι αναγνωρίζουμε ότι στον τομέα αυτών δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τόσες επενδύσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτή η μείωση. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν δεχόταν το στόχο αυτόν καθώς και το στόχο της μείωσης που θέσαμε για το 50 που θα ήταν ο πιο κοστολογικά αποτελεσματικός στόχος. Ας μιλήσω τώρα για το τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα. Τρεις, τρία συγκεκριμένα μέτρα που επεξεργάζονται η υπηρεσία μου. Πρώτον, οι θαλάσσιες εκπομπές η αύξηση των εκπομπών στον θαλάσσιο, το μέσο τομέα των θαλασσίων μεταφορών, υπονομεύει τις προσπάθειές μας να μειωθεί συνολικά οι εκπομπές, γιατί μεταξύ του 90 και του 7 η Ένωση συνολικά έχει μειώσει τις εκπομπές κατά 380, ε, εκατομμύρια τόνους, αλλά η αύξηση από την διακίνηση των πλοίων είναι 400 εκατομμύρια τόνοι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό αντισταθμίζει την μείωση. Και το χάσμα αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι εκπομπές από όλους τους τομείς της οικονομίας. Η οδηγία ETS έχει προβλέψει τα στοιχεία αυτά και άλλα στοιχεία δείχνουν ότι η ετήσια εξοικονόμηση καυσίμων θα μπορούσε να ανέλθει σε 125 δισεκατομμύρια δαλάρια. Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους τομείς της, ε, των μεταφορών μέσω εξοικονομήσεων ο Επίτροπος Μεταφορών και εγώ συναντηθήκαμε για τρίτη φορά με τους ενδιαφερόμενους στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών γιατί όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζήτησε αν δεν υπάρξει πρόοδος να έρθουν να μας κάνουν προτάσεις για του χρόνου. Και επομένως είχαμε τρεις σημαντικότατες και πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με υψηλού επίπεδου ενδιαφερομένους, εκπροσώπους δηλαδή των θαλασσίων μεταφορών και εκεί υπόθηκε ρητά ότι κάπου η αγορά κάνει κάτι λάθος. Εξετάζουμε λοιπόν την πιθανότητα να ληφθούν μέτρα εξοικονομήσεων ειδικά στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος το επόμενο έτος μέχρι να κάνουμε τις αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις πριν μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Αλλά σίγουρα εμείς προτιμούμε μια σφαιρική συνολική καθολική λύση. Δεύτερον, ετοιμάζουμε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το διοξίδιο του άνθρακος από αυτοκίνητα και φορτηγά η Λευκή Βίβλος σημειώνει ότι η αύξηση των εκπομπών από τους τρόπους αυτούς μεταφορών είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ήδη Έχουμε προβλέψει τον καθορισμό νέων στόχων για τις εκπομπές από τα νέου τύπου αυτοκίνητα που ήδη έχει αποδειχθεί ότι μειώνονται σε υψηλότερο ρυθμό από τότε που άρχισε να εφαρμο... άρχισαν να εφαρμόζονται τα νέα υποχρεωτικά κριτήρια για το διοξίδιο του άνθρακος. Μειώθηκαν κατά 20 γραμμάρια το χιλιόμετρο από τότε που υπάρχουν τα νέα αυτοκίνητα, ενώ στο παρελθόν ήταν μόνο 10 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Και η τάση αυτή αυξάνεται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία κάνει προσπάθεια, είναι στο σωστό δρόμο. Uh, Και για το 2020 ο στόχος μας είναι τα 25 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Βρίσκουμε ρεαλιστικό το στόχο αυτό γιατί και η βιομηχανία μας είπε ότι οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορέσουν να πετύχουν το στόχο αυτόν. Αυτό βέβαια είναι θετικό γιατί σημαίνει ότι όταν δοθεί η κατάλληλη όθηση προχωράνε τα πράγματα. Επίσης ζητήσατε να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε ως το τέλος του 12 να γίνει μία πρώτη αξιολόγηση για τα αυτοκίνητα. Άρχισε η μελέτη αυτή και τα αποτελέσματα θα αναφερθούν στις, στο τέλος του επόμενου έτους. Τρίτον, ετοιμάζουμε μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακος από βαρέα οχήματα υπολογίζεται ότι ευθύνονται για 66% των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Ένωση που ισοδυναμεί περίπου με το σύνολο των εκπομπών από αέριες και ποτάμιες μεταφορές. Είναι σημαντικό το ποσοστό λοιπόν. Αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για μεταφορά εμπορευμάτων και η μείωση των εκπομπών από βαρέα οχήματα είναι ένα από, τα βασικότερα, από τους βασικότερους μας στόχους γιατί θεωρούμε ότι θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη στρατηγική καταπολέμηση μείωση των συνολικών εκπομπών. Αν όμως και με τα βελτιωμένα αυτά βαρέα οχήματα συνεχίσουν οι εκπομπές, θα προετοιμάσουμε μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών και απολεοφορία, όχι μόνο από φορτηγά. Την έχουμε αρχίσει ήδη και θα την παρουσιάσουμε το 2013. Βεβαίως, ήδη αρχίσαμε διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. που την προσέχει και ιδιαίτερα και η διεθνής κοινότητα. Μιλάω για τις εναέριες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές. Η νομοθεσία αυτή εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο από το 8. Αλλά τρίτες χώρες με επικεφαλής στις Ηνωμένε Πολιτείες συνεχίζουν να πιέζουν την Ένωση για να μην εφαρμοστεί. Πρέπει όμως να σας πω ότι όλες οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες συμφωνούν, εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της νομοθεσίας αυτής. Μερικές φορές όταν ακούτε ορισμένες ακραίες δηλώσεις πρέπει να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα την εφαρμόζουν την νομοθεσία ό,τι και να λένε. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπήρξε μια υπόθεση προσφυγής Αμερικανικών εταιριών αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της απέρριψε, όλα τα αιτήματα των Αμερικανικών εταιριών. Δεν είναι αντίθετη η νομοθεσία με τους κανόνες της ΙΚΑΟ η οποία είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα είδος περιορισμού των εκπομπών και ο καλύτερος τρόπος θα ήταν μέσω των περιφερειακών συναλλαγών για τις εκπομπές. Δεν αντιτίθεται ούτε στη συνθήκη του Σικάγου, ούτε το UNFCC, ούτε υπάρχει θέμα ετεροδικίας, ούτε δεν δικαιολόγησε το δικαστήριο καμία από τις κατηγορίες που έθεσαν οι Ηνωμένε Πολιτείες. Στη νομική προσφυγή λοιπόν δεν δόθηκε δίκαιο. Και τώρα προσπαθούν να αυξήσουν την πολιτική τους πίεση. Εμείς ως Ένωση πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί σε αυτήν την νομοθεσία τονίζοντας ότι δεν έχουμε σκοπό να την αλλάξουμε πληροφορούμε τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις και υπήρξε στο Συμβούλιο υποστήριξη της θέσης αυτής. Στην τελευταία συνεδρία στη ΣΥΚΑΟ την περασμένη εβδομάδα η Ένωση επέδειξε ενωμένο μέτωπο για την υποστήριξη αυτής της νομοθεσίας. Πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι για πολλά χρόνια ζητούσαμε καθολική συνδυασμένη νομοθεσία για το θέμα της μείωσης των εκπομπών και τώρα αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε μέσω της συναλλαγής εκπομπών περιφερειακά, αντισταθμιστικά δηλαδή μέτρα. <coughs> Δεν είναι έκπληξη που ορισμένοι αντιτίθενται. Θα ήθελα όμως να σας αποσαφηνίσω μερικές λεπτομέρειες γιατί είμαι σίγουροι ότι σας θέτουν πολλά ερωτήματα οι πολίτες. Ένα, η αναλογικότητα. Στον τύπο βλέπετε συχνά αντιφατικά στοιχεία. Υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν στον αμερικανικό τύπο ότι κοστίζει 50 δολάρια παραπάνω κάθε ταξίδι για τα μέτρα αυτά. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μία πτήση Λονδίνο-Νέα Υόρκη αντιπροσωπεύει 1,5 ευρώ παραπάνω για τον κάθε επιβάτη. Φραγκφούρτη Πεκίνο 2 ευρώ παραπάνω. Μπορεί κανείς λοιπόν να πει ότι είναι γελιοδός χαμηλό το κόστος αυτό. Αλλά να ξέρουμε τα στοιχεία. Γιατί είναι τόσο χαμηλό το παραπάνω κόστος. Διότι στην νομοθεσία που εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο, 85% των συναλλαγών των αδειών εκπομπών που χορηγήθηκαν ήταν δωρεάν τον πρώτο χρόνο. Έχω ακούσει να λέγεται ότι θα είναι τεράστιο το πρόβλημα γιατί οι αεροπορικές εταιρείες θα πηγαίνουν, θα περνάνε από τα Ηνωμένα λέει Αραβικά λέει, Εμμυράτα λέει. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι μπορεί κάνει μια εταιρεία για να πάει από τη Φραγκφούρτη στο Πεκίνο για να εξοικονομήσει δύο ευρώ θα σταματήσει σε ενδιάμεσο σταθμό στα Εμμυράτα. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά έτσι είναι ότι αν τα εφαρμόζαμε μόνο για το δικό μας ένα χώρο, τότε πολλές εκπομπές αεροπορικές δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε καμία νομοθεσία, διότι μεγάλο τμήμα του εναερίου χώρου, το μεγαλύτερο, είναι πάνω από τη θάλασσα. Και θα βλέπατε τότε ότι οι αεροπορικές εταιρείε θα άρχιζαν να έχουν πολύ περίεργα δρομολόγια για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο και τα τρία θεσμικά όργανα δέχτηκαν την νομοθεσία ως έχει τέλος. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολύ καλό διάλογο με πολλές τρίτε χώρες για ισοδύναμα μέτρα. Δεν επιβάλλουμε σε κανέναν τι πρέπει να κάνει, αλλά προβλέπεται αν υπάρχουν αντισταθμιστικά ή ανάλογα μέτρα να βελτιώνεται έτσι ο διάλογος με τις τρίτες αυτές χώρες. Αν έχετε ισοδύναμα μέτρα τότε τα δεχόμαστε όσοι έχουν για να προσγειωθείτε στην Ευρώπη χωρίς πρόσθετο βάρος. Η Κίνα παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή εξετάζει το κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμόσει στόχους ανατομέα στις αεροπορικές της μεταφορές. Τέλος η Ένωση και θέλει και έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμοστεί ένα σφαιρικό καθολικό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές. Δυστυχώς η ΚΑΟ δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια και καλό θα ήταν να αρχίσει και εκείνη να το σκέφτεται το θέμα. Τέλος, για τρίτη φορά κύριε Πρόεδρε, οι υποδομές των εναερίων μεταφορών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτά τα ολοκληρωμένα δίκτυα για να επιτευχθούν οι κλιματολογικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης για το 20 για τη μείωση του ρόλου του διοξιδίου του άνθρακος στα καύσιμα και πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν όλα αυτά όχι μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές αλλά και για το συνδυασμό τους με τις υδροδρομικές και οδικές διάφτες. Πρέπει λοιπόν στον προϋπολογισμό μας να συμβάλλουμε στην απανθρακοποίηση των μεταφορών. Στο επόμενο MFF θα αναφέρουμε ότι πρέπει τουλάχιστον το 20% να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την γενικότερη στρατηγική του 2020, ιδιαίτερα για τη μετάβαση προς μια οικονομία με λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Να συνδυαστούν διάφοροι τρόποι μεταφορών για να διευκολυνθεί έτσι η μετάβαση από τις οδικές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στη δέσμη που προβλέψαμε είπαμε ότι η μετάβαση αυτή δεν σημαίνει να μειωθούν μόνο οι δημιουργίες νέων αυτοκινητοδρόμων, αλλά, α, αλλά λέγω και νέοι σιδηρόδρομοι. Όσο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, νομίζουμε ότι η μετάβαση αυτή θα βελτιώσει και τα δύο αυτά θέματα. Τέλος για τέταρτη φορά κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε εμείς στην Κομισιόν να γίνει ένας συνδυασμός των δικαιοδοσιών. Δεν μπορούμε να έχουμε χωριστά το σχεδιασμό, της μεταφορές, τις κλιματολογικές αλλαγές για την ανάπτυξη τελείως χωριστά. Όλα αυτά πρέπει να συνειδιαστούν παρά τον περιορισμό των πόρων που διαθέτουμε. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε αυτά και ελπίζω και το Κοινοβούλιο να δεχτεί το συνδυασμό αυτόν. Σας κατευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εγώ Επίτροπα. the... Και τώρα να περάσω στους συντονιστές. Έχουμε 35-40 λεπτά γιατί η Επιτροπός θα πρέπει να πάει στις 11.30 στην Επιτροπή Βιομηχανίας, άρα να είμαστε όσο το δυνατόν συντομότεροι και αν διαφωνείτε παρακαλώ βουλευτές με άλλους βουλευτές να μην ξεκινήσουμε κατεδίαν ζητήσει. Να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Γκρόσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Νομίζω ότι βρίσκεται σε μια επιτροπή η οποία αντιλαμβάνεται ότι οι μεταφορές από οικονομικής άποψης είναι πάρα πολύ σημαντικές, το οποίο ξεχνάμε πολύ και ότι φυσικά αποτελούν και μια μεγάλη πρόκληση για το περιβάλλον. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα μέτρα που υποστηρίξαμε, για παράδειγμα η Λευκή Βίβλος, επιδεικνύουν μια συνοχή και μία συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πτυχών που δεν θα πρέπει να είναι αντιφατική αλλά συμπληρωματική. Αλλά για να υπάρχει συμπληρωματικότητα χρειαζόμαστε κάποιους βασικούς κανόνες. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Να πω όμως το εξής. Η νομοθεσία και η κατεύθυνση που ακολουθούμε θα πρέπει όχι μόνο να αποφασίζεται αλλά και να εκτελείται να πραγματοποιείται κοιτώντα το λευκή βίβλο για το 2020, για το 2050 και κοιτώντα και τι έχει γίνει στο παρελθόν. Μερικοί από εμά ε, είχαν δει και τη λευκή βίβλο για το 2000. Αναρωτιόμαστε λοιπόν τι έγινε με τους στόχους που δεν πετύχαμε. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε τα μέσα για να ασκούμε την πολιτική αυτή, μεταξύ άλλων και τους χρηματοοικονομικούς πόρους και ο σχετικός φόρος αποτελεί σημαντική πτυχή που συνδέεται φυσικά και με την επικουρικότητα, αλλά και η υποστηρίξη σε έρευνα και ανάπτυξη. Και αν αντιληφθούμε τη σημασία στον τομέα του περιβάλλοντος, ε, του συνολικού πακέτου των μεταφορών και δούμε και το βάρος που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα, νομίζω ότι διαπιστώνουμε έλλειψη συνοχής. Τρίτον, είναι ακριβώς η συνοχή την οποία έδειξα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνοχή. Καταρχάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα παράδειγμα να δώσω. Στον τομέα του περιβάλλοντος θα μπορούσαμε να επενδύσουμε κατά την αρχή ο πληρώνει, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε earmarking. Ξέρετε τι δυσκολίες συμπεριλαμβάνεται το σύστημα αυτό στην εκτέλεσή του. Τα μέσα αυτά που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στον ε, τομέα των καθαρών μεταφορών. Αποτελεί θέμα σχεδόν ταμπού. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοχή, να πάρουμε το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Ήταν κάτι το οποίο γρήγορα, γρήγορα εφαρμόστηκε και σκοπό είχε εξοικονόμηση σχεδόν 20%. Νομίζω ότι αξίζει, επειδή μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις στο σημείο αυτό και δεν μιλάμε για μεγάλες μακροοικονομικές ε, αποφάσεις, αξίζει να ασκούμε μεγαλύτερη πίεση στον τομέα αυτό, γιατί πολύ γρήγορα μπορούμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνοχή και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. αλλά γίνονται διάφορες διασκέψεις και θα θέλαμε να ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον είναι εμ, αποφασιστική και ενιαία υποστήριξη στις πολιτικές αυτές. Δηλαδή, Αύριο θα υπάρχει ακόμα η ηλεκτρονική κινητικότητα ή μήπως θα υπάρχει πιθανότητα κάποιος ε, επιτρόπος για την ε, βιομηχανία να μην τον στηρίξει το θέμα αυτό και να αφαιθεί. Είναι λοιπόν μαζική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για να υπάρχει μια συνεκτική εικόνα και προς τα έξω. Γιατί ανησυχώ, και αυτό είναι το τελευταίο θέμα που θα θίξω, για το εξή. Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις και περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή ε, για να ανακύψουν προβλήματα και τελευταία στιγμή αλλάζουμε την απόψη μας και αναβάλουμε τη λήψη απόφασης όπως το ε, έγινε και στην περίπτωση των υγρών. Ίσως να μην το ξέρετε το θέμα αυτό, αλλά το είδαμε εδώ στην Επιτροπή. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας προβλέπεται για την τάδα νομοθεσία, για την τάδε ημερομηνία και τα κράτη-μέλη δεν θα θελήσουν να την εφαρμόσουν και μετά αποφασίστηκε μονομερός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει αναβολή της ε, ισχύω της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να το αποφύγουμε σε περίπτωση τέτοια σύγκρουση. και με την Αμερική αλλά και με άλλες χώρες. Θα πρέπει να το αποφύγουμε γιατί το θέμα εδώ πέρα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Αν σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα συμβαίνει, συμβεί κάτι τέτοιο εκ νέου, να σας πω ότι κάθε διμερή συζήτηση μεταξύ Ευρώπης και άλλων χωρών να τις ξεχάσετε, γιατί θα έχουμε αποτύχει. Δηλαδή, ποιο θα είναι το μήνυμα που θα στείλουμε, ότι κοιτάξτε, αν δεν θέλετε εσεί, εντάξει, θα αναθεωρήσουμε και εμεί τη θέση μα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σα παρακαλώ. Στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο να καταλάβετε ότι αν ακολουθήσετε τον δρόμο αυτό δεν θα υπάρχει περιθώριο επιστροφής. Ευχαριστώ για του σοσιαλιστέ ο κ. Ελκαντράουι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα ξεκινήσω και θα συμφωνήσω με τον Ματιό. Γιατί λέει ότι άλλο να αποφασίζουμε την νομοθεσία και άλλο να την εφαρμόζουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στον τομέα των μεταφορών που διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν, διστάζουν το λέω γενικά, να εφαρμόζουν συγκεκριμένα α, τμήματα της νομοθεσίας. Ε, το Single Sky αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε τεράστια ωφέλη να έχει για την Ευρώπη. Αλλά να ρωτήσω δύο πράγματα. Καταρχάς, αναφερθήκατε σε διάφορα συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες προτάσεις ε, τις οποίες θα καταθέσετε του επόμενου μήνες σε ό,τι αφορά κυρίως ε, την τυποποίηση του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά οχήματα. Πρόκειται για μέτρα τα οποία ασφαλώς θα αποδώσουν καρπούς. Ε, μιλήσατε ήδη και για τα ωφέλη που ήδη έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, ο δύσκολος τρόπος το μεγαλύτερο όφυλος θα πρέπει να το κερδίσουμε μακρυπρόθεσμα. Και αυτό θα έγκυται στην άλλη και διαφορετική χρήση των τομέων μεταφοράς. Αυτό το modal shift που πρέπει να γίνει για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς. Και αυτό θα προαπαιτήσει πιο βασικές και θεμελιώδες μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θεωρείτε ότι διαμορφώνεται και ο δικός σας ρόλος για να πετύχετε αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα. Στη Λευκή Βίβλο, την οποία μελετούμε, τη διαβάσαμε όλοι και συμφωνούμε με όλους αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους, όλα αυτά όμως αναφέρονται στο 2050. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε και πριν από το 2050 αποτελέσματα, να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αυτή η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση. Θα επανέλθω στο θέμα της ανταλλαγή ε, ρήπων για την αεροπορία. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την οποία και ψηφίσαμε. Νομίζω ότι νομικώς έχουμε δίκιο. Αυτό το υπογραμμίσατε άλλωστε κι εσείς λέτε ότι οι εταιρείε εντωμεταξύ σε προετοιμάζονται πλήρω. Αυτό φυσικά είναι θετικό νέο. Όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά, αλλά ξέρετε επίση ότι δεν υπάρχει πλέον νομικό θέμα. Το θέμα έχει καταστεί πολιτική φύση. Και άρα ερωτώ το εξή. Τώρα ε, απέχουμε δύο μήνε από την προθεσμία και ξέρετε ότι στο Αμερικανικό Κογκρέσο οι αντιδράσει είναι πολύ οξύε υπάρχουν απειλές με αντίπεινα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πώς αξιολογείτε λοιπόν αυτές τις απειλές. Πιστεύετε, ότι είναι απλά μια απειλή η οποία δεν θα εφαρμοστεί και αποτελεί απλά μέτρο πίεσης, μέσο ή προετοιμάσαστε ενδεχομένως και για πραγματική, ε, ένα πραγματικό πόλεμο εμπορικής φύσεως στο θέμα των αεροπορικών μεταφορών. Και τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει για να προτιμήσετε, για να προσπαθήσετε να πείσετε τα, τις τρίτες χώρες για αυτά που είπατε. Για το περιεχόμενο της νομοθεσίας και για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας. Επίση, τι σκέψεις έχουν γίνει σε πολιτικό επίπεδο για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένη τέτοια κατάσταση. Και αν το πρόβλημα δεν πάυσει, πώς θα αντιδράσετε από αρχή του επόμενου έτους. Thank Σας ευχαριστώ, η κυρία Μάισνερ, για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την Επίτροπο. Έχετε φυσικά δίκιο. Να ξεκινήσω λέγοντας αυτό δεν μπορούμε να τα κοιτάζουμε όλα κατακαιρματισμένα, παραγωγή, μεταφορές, περιβάλλον, όλα αυτά θα πρέπει να ειδωθούν σε ένα σύνολο. Αυτό καμιά φορά είναι δύσκολο, αλλά στην τελική ανάλυση, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους για το περιβάλλον, θα πρέπει σε όλους τους πολιτικούς τομείς να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι μεταφορές, το είπε ο Ματιό Γκρός, για την ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε όλα τα μέσα μεταφοράς, αυτό πρέπει να το τονίζουμε για τη διαφορετική και η περιβαλλοντική φιλικότητα των διάφορων τομέων μεταφοράς και σε όλους τους τομείς θα πρέπει να δράσουμε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αλλά και σε ό,τι αφορά την παραγωγή, για παράδειγμα. Γιατί πολλά πετυχαίνουμε στα υλικά, για παράδειγμα των κατασκευών. Υπάρχουν νέα υλικά για αεροπλάνα, για αυτοκίνητα. Τα αεροπλάνα κατασκευάζονται προκειμένου να είναι πιο ελαφριά, προκειμένου να χρησιμοποιούν λιγότερο καύσιμο όταν χρησιμοποιούνται. Πολλά λοιπόν γίνονται, αναζητώνται εναλλακτικά καύσιμα. Για παράδειγμα, ε, για τα πλοία χρησιμοποιούνται διάφορες, ε, διάφοροι μηχανισμοί κίνησης, ανεξάρτητα μάλλον, ανάλογα με το αν ε, κινούνται κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα ή σε Άρα πολλά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στα πλοία πάλι για παράδειγμα. Υπάρχουν ε, πλοία ουδέτερα ως προς τις εκπομπές. Αλλά χρειάζονται και μια σχετική υποδομία. Το υποδομή. Το υγροποιημένο αέριο αποτελεί επίσης ένα ζήτημα σημαντικό. αυτά γενικά. Όντω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν διάφορους τομείς. Το κάνετε άλλωστε. Είπατε ότι χρειαζόμαστε μια πολυμερή προσέγγιση, προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πολιτική αυτή. Δύο θέματα να θίξω για τα ευφυή e συστήματα μεταφορών. Μπορούν να βοηθήσουν πολύ για την ε, αποτελεσματική διαμόρφωση των μεταφορών και για την καταπολέμηση την πρόληψη, αν θέλετε, δημιουργίας ε, εκπομπών. Χρειαζόμαστε φυσικά μέσα για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, αυτοκινητόδρομοι που έχουν δημιουργηθεί για την πρόληψη των μποτιλιαρισμάτων. Ρωτώ λοιπόν για τις αερομεταφορές. Είναι ασφαλώς καθήκον της ΙΚΑΟ να φροντίζει για την ε, εκπομπή λιγότερων ρήπων. Τι θέλει η Ευρώπη σήμερα, κάτι πολύ ορθό. Να υπάρχει α, σύστημα ανταλλαγή ρήπων και για τις αερομεταφορές. Αλλά υπάρχει σχετική σύμβαση στη Γερμανία ότι αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τι θα γίνει λοιπόν αν ε, η Κίνα ορίσει ότι θα υπάρχουν κυρώσει για τις ευρωπαϊκές εταιρείε ή αν η ΕΠΑ δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει. Τι δυνατότητε θα έχετε να αντιδράσετε στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και την Επιτροπή. Καλό είναι που ακούμε από πλευρά των ε, προγραμμάτων ε, υποδομής υποστήριξη για project όπως το Caesar, το Caesar. Εγώ συνεργάστηκα και με τους συναδέλφους που ασχολούνται με υποδομές διαστήματος για τις μεταφορές. Δεν έχουμε όλοι πάρα πολύ χρόνο για να μιλήσουμε, αλλά να επικεντρωθώ στο σύστημα εμπορίας ρήπων. Να είμαι ειλικρινής, κυρία η κυρία Χέντεγκαρτ δεν ήταν εδώ όταν εισήχθη το σύστημα αυτό. Και ανησυχώ για το εξή. Ήμουν εκτός του κοινοβουλίου. Δούλευα στον ιδιωτικό κλάδο. Και όταν ξεκίνησε η εισαγωγή του της αεροπορίας στο σύστημα αυτό, πολλέ πηγές κατέστησαν σαφέ ότι θα ήταν τεράστιε οι δυσκολίες, γιατί πολύ απλά πρόκειται για φορολογία. Δεν πρόκειται για τέλο, πρόκειται για φορολογία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αρμοδιότητα να φορολογούμε εταιρείε άλλων χωρών, τρίτων χωρών. Και τώρα κανείς δεν εκπλήσεται. Και εγώ όταν ε, βρέθηκα για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, γιατί το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αμερική. Η Επιτροπή κατέθεσε την ε, πρόταση και 160 χώρες έγραψαν επιστολές ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας προβλήματα που είχαν. Αγνοήθηκαν. Αγνοήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Άρα πολύ λυπάμαι κυρία Χέντεγκάρτ. Μας εξηγήσατε με πολύ καλό τρόπο πόσο φρικτή είναι οι Αμερικανοί που δεν μας ακούν, αλλά δεν ξέρω να υπήρξε κανένας στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος που να εκπλήχθηκε από το γεγονός αυτό. Γιατί προσπαθείτε να αποτρέψετε τον απότρεπτο. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα... Έχετε φτάσει σε ένα σημείο που πιστεύετε την ίδια σας την προπαγάνδα. Δεν είμαστε σε θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προδιαγράψουμε στον άλλο κόσμο τι θα πρέπει να κάνει. Γιατί όταν θα τεθούν ισότιμα μέτρα, ποιο θα το αποφασίσει, εσεί θα το αποφασίσετε, αν εκείνη ναι. βγήκε και πει ότι έβγαλε εγώ ένα ισοδύναμο μέτρο. Και τελικά, τι θα πούμε ότι α, το ένα μα αρέσει, το άλλο δεν μα αρέσει. Και τελικά, πού μένουμε. Γιατί το θέμα αυτό δεν, είναι, δεν αφορά μόνο την Αμερική. Και αν ε, έχετε συνομιλήσει με κάποιους από την Κίνα και θεωρείτε ότι είναι σχετικά ε, ήπια αντίδραση, να σας πω ότι δεν είναι ήπια η αντίδραση ούτε της Κίνας, ούτε της Ρωσίας, ούτε τον ΗΠΑ. Μπορεί να μην σας το λένε κατά πρόσωπο, αλλά σίγουρα δεν κρύβουν την ε, αντίδρασή τους. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά μη δημοφιλές μέτρο και θεωρώ ότι είναι και άδικο, γιατί δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει με συλλογή φόρων. Εγώ δεν ε, έχω πρόβλημα να εισάγουμε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ρήπανση. Αλλά αυτό ποτέ δεν ήταν ο στόχος μας. Άλλο να έχουμε ένα σύστημα ανταλλαγής ρήπων, άμεσο, αλλά αυτό δεν, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το σύστημα. Και θα κλείσω στο σημείο αυτό, Πρόεδρε, λέγοντας είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ θα εκπροσωπήσω και τους, ε, τις επιχειρήσεις και τις εταιρείε του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί όταν το σύστημα αυτό ξεκινήσει τον Ιανουάριο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αν κανείς θα πληρώσει ή όχι, γιατί να υποστηρίξω ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα εφαρμόσει και θα επιβάλλει πιο πολλή φορολογία στις επιχειρήσεις μου που προσπαθούν να τα επεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της αλυσίδας, από τον τουρισμό, από τις κατασκευαστικές, από τις ε, αεροπορικές δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πετύχει. Προσπαθήστε να, προσπαθείτε να ανοίξετε τα σχήρα σα και να πείτε ότι θα λειτουργήσει το σύστημα. Θα ήθελα όμω να ξέρω ποιο είναι το εναλλακτικό σα σχέδιο, Επιτροπέ. Άμα. Ο κύριο Κράμερ. Να σα ευχαριστήσω και για την παρουσίαση. Θα ήθελα να υποστηρίξω την αντίθεση θέση. Έχετε όμω δίκιο σε ένα σημείο, κυρία Φώσταρ. Το θέμα είναι η φορολογική νομοθεσία και σε ό,τι αφορά τι αερομεταφορέ είναι πραγματικά μη κοινωνική και απαράδεκτη η φορολογία, γιατί ο Ευρωπαίος φορολογούμενος κάθε χρόνο πληρώνει 30 δισεκατομμύρια ευρώ στις ε, αεροπορικές, γιατί δεν ε, πληρώνουν φόρο επί της κυροζήνης. Και αυτό δεν το πληρώνει μια-δυο φορές όταν πετάει. Όχι. Αυτό ευνοεί αυτούς που πετάνε πολύ και που έχουν πολλά χρήματα στα τελική ανάλυση και το σύστημα ανταλλαγής ρήπων έγινε αποδεκτό από τις εταιρείε γιατί ξέραν ότι αν δεν το δεχόντουσαν θα είχαν ένα ευρώ φορολογία για την κυροζήνη. Αν προκύψει λοιπόν αυτή η αντίδραση, μπορείτε να τους αντιπροτείνετε να πληρώσουν φόρο επί της κυροζήνης, γιατί η συνθήκη για το, του Σικάγο περιλαμβάνει και λέει ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί η κεροζίνη όταν έρχεται ένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να φορολογηθεί η κυριοζήνη που α, βάζει ένα αεροπλάνο, για παράδειγμα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και νομίζω ότι αν ατεθεί αυτό ω εναλλακτική λύση, θα σιωπήσουν οι ευρωπαϊκέ όλε οι εταιρείε όλου του κόσμου, οι αεροπορικέ, γιατί πολύ απλά είναι πιο ακριβό το σύστημα αυτό αλλά μετά τις αρνητικές ε, εμπειρίες με τις ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες τότε αντιστάθηκαν, εγώ θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Η προνομιακή αυτή μεταχείριση των αεροπορικών επιχειρήσεων θα συνεχίσει να υπάρχει και θα πρέπει να, να αλλάξει. Είπατε, δεν μπορούμε να έχουμε από πλευρά. Ε, δεν μπορούμε να ασκούμε πολιτική για το περιβάλλον και για τι μεταφορέ και να θεωρούμε ότι δεν συνδέονται. Αλλά δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώ και στην Ευρώπη δεν συνδέονται. Και φυσικά αυτό που κυριαρχεί είναι το χρήμα και ξέρουμε που πάει το χρήμα. 60% πάει στα, στο, στις οδικές μεταφορές, 20% πάει στους σιδηροδρόμους. Ξέρουμε που πάνε τα χρήματα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να είναι αντίθετη αυτή η ισορροπία. Κοιτώντα για τα μεγάλα project, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μεγάλες, ε, μάλλον ε, την ε, συνδρομική γραμμή Ulm Ulm-Stuttgart και χρησιμοποιείται μάλλον κατασκευάζεται μια νέα γραμμή τριών δισεκατομμυρίων, η οποία όμως και αυτή δεν είναι κατάλληλη για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Βερολίνου και Μπρέσλαου. Οικοδομείται άλλη γραμμή. Μα θα πρέπει να επένδεται προκειμένου οι επενδύσεις με το μεγαλύτερο όφελος να προωθηθούν. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω για την ηχορύπανση. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα αν επενδύσουμε στα σχετικά υλικά. Αλλά αυτό απαγορεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση. Με τα μισά χρήματα θα μπορούσαμε στα 10 χρόνια να μειώσουμε το, την ηχορύπανση κατά το ίμιση στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Με 4,5 δις από, και όχι με 10 με τα μεγάλα project στον Δούναβη. Επενδύουμε ε, σε μεγάλα project όπου, από όπου περνάνε ένα-δύο πλοία κάθε μέρα. Στη Γερμανία 40 δισεκατομμύρια επενδύσαμε τα τελευταία χρόνια στο συνδρομικό δίκτυο και διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί 20% το επιβατικό κοινό. Δηλαδή δεν επενδύουμε εκεί που πραγματικά θα έπρεπε να επενδύουμε. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην προστασία του κλίματος, γιατί δεν έχουμε εναλλακτική. Τελευταίο σημείο. Είπατε ότι η βιομηχανία τα πηγαίνει πιο γρήγορα ε, μάλλον καταφέρει πιο πολλά αποτελέσματα και πιο γρήγορα αποτελέσματα για τη μείωση των εκπομπών στα αυτοκίνητα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό δεν είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν θα πρέπει να ακούμε πάντα και τα παράπονα της ε, βιομηχανίας, αλλά είναι ντροπή να τα πηγαίνει πιο γρήγορα η βιομηχανία από τους δικούς μας τους στόχους. Και τελευταίο τελευταίο, είπατε ότι οι εκπομπές για τα αυτοκίνητα έχουν μειωθεί. όντω αλλά φυσικά σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυξηθεί, γιατί η μείωση απορροφάται και αντισταθμίζεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων. Αυτό το επιβεβαιώνεται ή όχι. Thank τελείωσαν οι εκπρόσωποι των ομάδων. Παρακαλώ τους συναδέλφους να είναι πολύ συγκεκριμένοι. Κυρία Ντεβεράκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μόνο μερικά για την οδηγία ΤΕΣΕ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία 90% τον ε, Ιούνιο του 2008 και αποτελεί σταθμό για την ε, περιβαλλοντική πολιτική. Μετά από μερικές εβδομάδες ε, θέσεις σε ισχύ αυτών των μέτρων, οι χώρες αρχίζουν και ξυπνούν η μία μετά την άλλη και η δήλωση του Συμβουλίου της ΟΑΣΕΗ στις 2 ε, Νοεμβρίου ε, δείχνει ότι υπάρχει πλήρης άγνοια των μέτρων που προτείνονται από αυτήν την οδηγία. Υπάρχει από τη μια ο κανόνας de minimis όπου εξαιρούνται καμιά εκατοσταριά χώρες από αυτήν την οδηγία και το άρθρο 100β της οδηγίας ε, για τις τρίτες χώρες οι οποίες ε, θα αναλάβουν ε, ισοδύναμα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν χρειάζεται εξήγηση και, πυθ... και πυθός. Πρέπει λοιπόν εμείς ε, να ενισχύσουμε τον διάλογο με τις τρίτες χώρες για να βρούμε μια γρήγορη και διαπραγματευμένη λύση και να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο ε, ζημιογόνων αντιπίνων για τις αεροπορικές μας εταιρείες. Θα πρέπει εμείς όμως να σταθούμε σταθεροί στις θέσεις μας γιατί πρέπει να προασπιστούμε τις αποφάσεις μας. Ελπίζω σε μερικούς μήνες ε, να είμαστε ιδιαίτερα, να εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη θέση σε ισχύ της οδηγίας ΤΕΕΣ και η Κομισιόν να έχει πετύχει το παιχνίδι της πυθούς έναντι των εταίρων μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω σε ποια εναλλακτική πραγματικότητα ζείτε κυρία Επίτροπε. Μάθατε ότι υπάρχει μια σοβαρή παγκόσμια κρίση. που εστιάζεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ με αυτά που είπατε σήμερα ζητάτε όλο και περισσότερη διευθέτηση, περισσότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, κινδύνους για την απασχόληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναγνωρίζετε καθόλου την κρίση σε αυτά που είπατε. Η κυρία Φώστερ κάλυψε το θέμα του συστήματος ETS στις αεροπορικές μεταφορές, αλλά υπάρχουν και δύο άλλοι τομείς. Οι θαλάσσιες εκπομπές όπου φαντάζομαι ότι μιλήσατε με σφαιρικά στοιχεία. Αν αυξάνονται σφαιρικά οι εκπομπές εκεί και θέλουμε να μειωθούν, τότε βεβαίως χρειαζόμαστε σφαιρικές λύσεις, σαν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίσουμε με το ζόρι να εφαρμόζουμε εθελοντικά και μονομερός τέτοια μέτρα, τότε όλο και περισσότερες εταιρείες και θα μετεκατασταθούν εκτός Ένωσης. Εγώ δεν είμαι κατά της σύναψης σφαιρικών συμφωνιών περιορισμού αλλά να βάζουμε την Ευρώπη σε ανταγωνιστικά υποδεέστερη θέση είναι παράλογο. Δεύτερον, το θέμα των οδικών μεταφαρών. Εγώ εκπροσωπώ μια περιφέρεια που βρίσκεται στο κέντρο του οδικού συστήματος του ΙΤΑΒ. Πάνω από 900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών εδράζονται στην περιφέρειά μου. Και πριν από μερικά χρόνια έκανα μια μελέτη που έδειξε ότι αυτό που δεν θα ήθελαν ούτε από την Εθνική Κυβέρνηση ούτε από την Ένωση ήταν παραπάνω νομοθεσία γιατί ήδη αγωνίζονται για να επιβιώσουν και ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε σήμερα κυρία Επίτροπε σημαίνει ότι θα φαλιρίσουν και θα δημιουργηθεί επομένως περισσότερη ανεργία εκεί και αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε η κυρία Ντουράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητά σας κύριε Επίτροπε για το ΕΤΕΣ. Και θέλω να διορθώσω κάτι για το, το οποίο υπόθηκε για ένα προηγούμενο ντοσιέ ε, που αντιπαρέτεθε την Ευρώπη κατά τον ΙΠΑ ήταν το περίφημο ε, το Αλικάο ήταν το περίφημο κίτ ε, κατά του θορύβου τότε έλεγε η Αμερική ότι θα έπρεπε να ε, ε, ξαναδώσουμε άδειες, να ελέγξουμε τα παλιά αεροπλάνα και να τα αφήσουμε να πετάνε. Σήμερα όμως έχουμε μία απόφαση του δικαστηρίου που μας δίνει δίκιο, όπου σήμερα δεν έχουμε κανένα λόγο να ε, κατεβάσουμε τα στάνταρ μας και οι απειλές δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζουν και μετά αν υπάρξει προσφυγή τότε να οργανώσουμε μια διαιτησία. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα αναφέρατε για τις δεσμευτικές νομοθεσίες που έχουν αποτέλεσμα, για τις αναγκαστικές νομοθεσίες που έχουν αποτέλεσμα ε, και στην βιομηχανία, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι θα ήταν ένας δραστικός τρόπος άμα Άμα η βιομηχανία έφτιαχνε αυτοκίνητα ε, με, λιγότερο, με μικρότερο κυβισμό και με λιγότερες δυνατότητες να τρέχουν τόσο γρήγορα. Ταυτόχρονα δημιουργώντας κίνητρα για την ε, κινητικότητα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Κόκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την ε, εργασία της και έχω μία ερώτηση. Καταλήξατε σε συμφωνία με τους άλλους επιτρόπους ε, για τα οικονομικά μέτρα έναντι της οικονομικής και πολιτικής ε, κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι σήμερα ε, δόθηκε μία προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος ύφεσης. Τα μέτρα τα οποία όμως εσείς ε, λαμβάνετε για το 2003 είναι μέτρα κατά της ύφεσης. Προβλέπετε επίσης να μειώσετε τις εκπομπές ε, για τα αυτοκίνητα μέχρι το 2013. Ευχαριστώ κύριε Κόχ. Και εγώ να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Πριν έρθω στην αεροπορία να αναφέρω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καταρχήν έγινε λόγος για τις θαλάσσιες μεταφορές. Πράγματι, το καλοκαίρι πετύχαμε στη Διεθνή Οργάνωση Θαλασσίων Μεταφορών να δημιουργηθεί ένας πίνακας, ένας δείκτης των εκπομπών τους. Και πώς το πετύχαμε αυτό, Α, κυρίως από την πίεση της Ένωσης είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να επιτευχθεί η διεθνής πρόοδος. Ο κύριος Γκραντς αναφέρθηκε στο θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας. Όταν συναντήθηκε η Κομισιόν με προέδρους επιτροπών, ο κύριος Σίμψον μας το ξεκαθάρισε αυτό το θέμα ότι χρειάζεται σωστή εφαρμογή Όλοι και οι χώρες μέλη και οι Κομισιόν πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Τέλος, για την έρευνα πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτή την εποχή της λιτότητας δεν είναι τυχαίο ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές που δημοσιεύσαμε δίνανε περισσότερα χρήματα μόνο στην έρευνα. Από 50 κάτι δισεκατομμύρια σε 80. Όχι μόνο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των καυσίμων, αλλά και γενικότερα γιατί αν ακούσουμε πόσες ιδέες έχουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για την βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών, για την επίλυση του α ή του β προβλήματος που αντιμετωπίζουν πράγματι στη ζωή τους, βλέπουμε ότι είναι κάτι που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικότερα. Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία. Μιλήσατε για έξυπνη διαχείριση των μεταφορών ναι. Αντί να πληρώνουμε για την κατασκευή όλο και περισσότερων αυτοκινητοδρόμων ή διαδρόμων τους, θα έπρεπε να κατανείμουμε καλύτερα τις μεταφορές και να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες υποδομές πιο ελαστικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Είναι κάτι ανάλογο με την οδηγία Open Skies. και είναι και κάτι που το καταλαβαίνουν εύκολα και οι εκλογείς και οι πολίτες. Μπορούν να εξοικονομηθούν πολλές εκπομπές και χρήματα και χρόνος απλώς και μόνο μέσω της καλύτερης χρησιμοποίησης των υποδομών που διαθέτουμε και της οργάνωσης. Και τώρα για τις ε, αεραπορικές μεταφορές. και για το αν ξέρω ότι υπάρχει κρίση. Αν ήθελα να είμαι και εγώ τόσο ομός όσο ο κύριος Μπλακμπον θα σας έλεγα ότι ούτε από εσά άκουσα να λέτε τίποτα για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η σφαιρική συμφωνία που ζητάτε. Το σκεφτήκαμε πολλά χρόνια, προσπαθήσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε. Και ακόμη το προσπαθούμε Η Ευρώπη θέλει να υπάρξει πρόοδος για μια σφαιρική διευθέτηση του προβλήματος των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών. Προσπαθούμε να το πετύχουμε. Αλλά επίσης από εδώ ακούστηκε ένα θέμα, ένα ερώτημα για την κρίση στην Κομισιόν. εξετάζουμε πολύ σοβαρά όχι μόνο πώς να αντιμετωπιστεί η κρίση αλλά και πώς να αναπτυχθεί στρατηγική για να βγει η Ευρώπη από την κρίση. Γιατί δεν έχουμε μόνο χρηματοπιστωτική κρίση, έχουμε μια πολύ δομικότερη κρίση. Δημόσια συστήματα πολύ, με πολλές δαπάνες, με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα κλπ. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων και ενεργείας. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων για χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας κτλ. από όπου αγοράζουμε όλο και ακριβότερο πετρέλαιο και αέριο. Είναι αυτό όφρον να φεύγουν χρήματα από την Ευρώπη αντί να επενδύονται σε πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας μέσα στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι αν επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές με καλύτερους μετρητές, συστήματα διανομής, καλύτερο σιδηρόδρομο, πιο ενεργειακά αποτελεσματικά κτίρια, τότε θα μπορούσε να φανεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όχι μόνο για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλες χώρες αλλά και για να επενδύσουμε στις χώρες μας να δημιουργήσουμε χώρες, ε, θέσεις απασχόλησης. Καλύτερα δίκτυα συγκοινωνιών ή ενεργειακής διανομής. Και δεν θα το κάνουν αυτό οι Κινέζοι, εμείς θα το κάνουμε. Γι' αυτό αυτόν τον τρόπο θεωρούμε σαν έναν τρόπο έξοδο από την κρίση. Δεν είναι ο μόνος βέβαια. Αλλά αφού υπάρχει όλο και περισσότερη ανταγωνιστικότητα, πρέπει και εμείς να δούμε στο θέμα ας πούμε των ανανεωσίμων και βιωσιμότερων πηγών ενεργείας, ότι θα μπορούσαμε και εμείς σε αυτό να είμαστε ανταγωνιστικότεροι. Τέλος, είδαμε ότι από το 8 μέχρι το 10 ο τομέας της ενεργειακής εξοικονόμησης δημιούργησε θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό λέμε ότι το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών της αντιμετώπισης τους είναι θέμα αποτελεσματικότερη χρήση ενεργείας που να γίνει και κίνητρο δημιουργία θέσεων Απασχόληση. Τέλος, για αυτό το τελευταίο θέμα θα ήθελα να πω απλώς ότι κατανοώ ότι ορισμένοι διαφωνούν. Εγώ όμως ως Επίτροπος Κλιματολογικών Αλλαγών κληρονόμησα ένα νομοθέτημα με σύμφωνη γνώμη και του Κοινοβουλίου και είτε ψηφίσατε υπέρ είτε κατά του νομοθετήματος αυτού, όλοι οι Ευρωπαίοι θα δεχόταν ότι δεν θα ήταν φρόνιμο η Κίνα να εμφαίνεται στους Financial Times να λέει αν η Ευρώπη δεν αλλάξει <coughs> την νομοθεσία της τότε θα πάρουμε μέτρα κατά του Ερμπάς και τα λοιπά. Όταν βλέπουμε τέτοιους τίτλους πώς αντιδρούμε, αλλάζουμε την νομοθεσία μας επειδή το είπε η Κίνα. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Σας ευχαριστώ για, όλα τα καλά σας λόγια. Εμείς κάνουμε πολλές διαβουλεύσεις. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στη Μόσχα όπου και πριν από δύο εβδομάδες στην Κίνα. Να ξέρετε λοιπόν να είστε βέβαιοι ότι και οι αντιπροσωπείες μας τα λένε αυτά σε όλο τον κόσμο. Είναι όμως πολύ σημαντικό και οι εκλελεγμένοι εκπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζουν ότι πρέπει να υποστηρίζουν αυτή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι συμφέρον τους. Η κυρία Ντουράν είπε ότι μερικές χώρες διαμαρτύρονται και ξερούνται από την νομοθεσία αυτή, αλλά και οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες δεν συμμετέχουν γιατί δεν έχουν αρκετές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα όπως τα είπατε. Τέλος, δεν πρόκειται για φόρο. Είναι λάθος να λέμε ότι είναι φόρος. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν είναι φόρος και το ξεκαθάρισε και το δικαστήριο. Δεν είναι φόρος. Οι φόροι για, τα... για τους αερολιμένες και λοιπά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ στόχος μας είναι να δημιουργηθεί κίνητρο για τις αεροπορικές μεταφορές ώστε να είναι οι εταιρείε να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά αεροπλάνα, αποτελεσματικότερη χρήση καυσίμων αν ανανεώνουν το στόχο τους να πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα αεροπλάνα και να είναι πιο αποτελεσματική και οικονομική και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσβίωση, η απογείωση κλπ. Τέλος, για άλλους τομείς τα έχουμε κάνει αυτά. Τομείς που εκτίθενται άμεσα στην, στον ανταγωνισμό. Και ο λόγος για τον οποίο η αεροπορία συμπεριλήφθηκε ήταν ότι πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς που διαθέτουμε που είναι πράγματι παγκόσμιας σημασίας δεν μπορούμε να στέλνουμε το λογαριασμό των μέτρων μας μόνο στους μεταποιητές και στους υπόλοιπους βιομήχανες ή στους πελάτες, αλλά πρέπει και στους επιβάτες και επιβάτριες. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε στενά με πολλές χώρες για να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, αλλά αυτό το εναλλακτικό σχέδιο που είπατε, εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε νυφάλιοι, να συνεργαστούμε με όλους μας τους εταίρους, να ψάξουμε λύσεις και μην πιστεύετε ότι την 1η Ιανουαρίου αρχίζουν οι διαμάχες. Όχι θα δοθούν εξαιρέσει, άδειε, δεν ξέρουμε πόσες για κάθε εταιρεία, για τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Και μόνο το 13 θα γίνει το πραγματικό επόμενο βήμα. Μη φοβάστε λοιπόν, δεν πρόκειται την πρωτοχρονιά να αρχίσουν τα προβλήματα και οι διαμάχες. Αλλά σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την προσοχή σας και την ειλικρινή σας συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Χέντεγκάρτ. θα πάτε τώρα αλλού μας είπατε. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία συνάδελφοι και συναδελφέ. Τώρα λίγη η συνεδρίαση. Η επόμενη μας συνεδρίαση Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού είναι 21η Νοεμβρίου Δευτέρα στις 3 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ τους ερμηνευτάς και τις ερμηνεύτριες. Λίγη συνεδρίαση.